καλημέρα σας. επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν ε, διανεμηθεί και διατίθεται. έχετε αντιρρήσεις; όχι από ό,τι βλέπω. οπότε και εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά. Ε, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει στείλει ένα αίτημα διορισμού ε, σε ε, επιτροπή που επισυνάπτεται στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και αν δεν διαφωνήσει κανείς ε, θεωρείται αυτός ο διορισμός εγκεκριμένος. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα στην διάταξη Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Υπάτη Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την κατάσταση στη Συρία. Σε εκπροσώπηση της Αντιπροέδρου και υπάτης εκπροσώπου θα πάρει το λόγο ο κύριος Ιωάννης Χάν. Παρακαλώ κύριε Επιτροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πόλεμος στη Συρία έχει μπει σε νέα φάση, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων ε, Πολιτειών ότι θα αποσύρουν <clears throat> τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ωστόσο, η πολιτική λύση δεν διαφαίνεται ακόμα. Ο μόνος βιώσιμος τρόπος να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι μια λύση με διαπραγματεύσει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε μια διχοτόμηση της Συρίας δεν πρόκειται να βοηθήσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της στη χώρα ούτε στην περιοχή. Η βορειοανατολική Συρία ε, τώρα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων ε, του καθεστώτος των ΗΠΑ, της ε, Τουρκίας, της Ρωσίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Δεν έχει ιτηθεί κατά κράτος το Ισλαμικό κράτος και μπορεί να επανέλθει στη συνέχεια. Κατανοούμε τις ανησυχίες της Τουρκίας, αλλά αυτό μπορεί μόνο ε, να λυθεί εφόσον διαφυλαχθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ακαιρεότητα ε, της Συρίας. Θα πρέπει να προστατεύονται όλες οι εθνότητες, ε, όλες οι θρησκείες και να αποφεύγονται νέα δεινά και συγκρούσεις. Στο μεταξύ, η Αλκάιντα στη Συρία, που προηγουμένως λεγόταν HDS ή Αλνούστρα, ε, εξακολουθεί να ελέγχει το Ιντλίμπ και τη γύρω περιοχή. Γι' αυτό ε, ως μέτρο προφύλαξης ε, δεν συνεχίζονται οι ε, επιχειρήσεις όπως και στο Νότο. Ε, είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Το μόνο θετικό είναι ότι έχει φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια ε, στα σύνορα με την Ιορδανία, στον καταβλισμό Ράκπαν, όπου ε, διαμένουν 60.000 Σύριοι, άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια παντού. Ε, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα σύνορα ε, και όλες οι ε, διαβάσεις και στη βορειοανατολική και στη βορειοδυτική Σύρια. Ιδιαίτερα τώρα που είναι χειμώνας και έχουμε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και πολλά παιδιά μεταξύ αυτών και αγωνίζονται να επιβιώσουν. Θα εξακολουθούμε να προστατεύουμε τους αμάχους σε οποιαδήποτε επίθεση και στοχεύουμε και στην προστασία των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκεί όχι στις αυθαίρετες ε, συλλήψεις και την ε, αναγκαστική στράτευση. Ε, η διαφθορά και η οικονομία του πολέμου παραμένουν οι μόνοι πηγή εσόδων και διαβίωσης για κάποιους ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς άλλος δεν μπορεί να βοηθήσει την ανοικοδόμηση εφόσον δεν υπάρξει πολιτική συμφωνία και ενώ, το καθεστώς δεν συμμορφώνεται ε, με τις αποφάσεις του ΕΕ και δεν βελτιώνει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα. Είπα η αρμοστία εξακολουθεί να μας λέει ότι οι ε, προϋποθέσεις για επαναπατρισμό ε, με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και μονιμότητα δεν είναι ακόμα δεδομένες για τους επαναπατριζομένους θα πρέπει να υπάρξουν οι σωστές και απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους Σύρους να γυρίσουν σε μια χώρα όπου κινδυνεύουν να τους συλλάβουν αυθαίρετα, να τους στρατολογήσουν αναγκαστικά και ακόμα και να τους βασανίσουν. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την πολιτική διαδικασία στη Γενέβη ε, ως τη μόνη ρεαλιστική λύση. Δεν μπορούμε, ε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παγώσουμε τη σύραξη εκεί. Αυτό θα σημαίνει περισσότερα δεινά, περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση, περισσότερη αστάθεια στην περιοχή και περισσότερη βία. Η κυρία Μογκερίνη είναι σε στενή ε, συνεργασία με τον κύριο Πέτερσον που είναι ε, ειδικό εντεταλμένος του ΟΗΕ. Επίσης ε, προσπαθεί να λανσάρει ε, και πάλι τη διαδικασία της Γενέβης. Για να γίνει αυτό, στα μέσα Μαρτίου θα φιλοξενήσουμε ε, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη μια διάσκεψη στι Βρυξέλλε που θα βασιστεί σε τρει πυλώνε. Υποστήριξη τη πολιτική διαδικασία, ανθρωπιστική βοήθεια και ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχο μα θα είναι να εξασφαλίσουμε υποσχέσεις ε, δωρεών για να αντιμετωπιστούν οι μόνιμε πάγιε ανάγκε των σύρων και των χωρών που έχουν υποδεχθεί τόσου πολλού πρόσφυγε. Φέτο επίση θα υποδεχθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι Βρυξέλλε μια ημέρα διαλόγου με υπουργού, και εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών από τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία. Ο λαός της Συρίας ζητάει μόνιμη, βιώσιμη λύση στον πόλεμο. Ζητούν μια χώρα όπου κάθε Σύρος να έχει τη θέση του παρόλες τις διαφορές ε, εθνότητας, θρησκευτικέ, πολιτικές και κοινωνικού ε, υποβάθρο προέλευση. Ε, τους αξίζει μια πολιτική λύση που θα οδηγήσει στη συμφιλίωση, στη ρανικοδόμηση και σε μια δημοκρατική Σύρια χωρίς αποκλεισμού. Αυτό εξακολουθεί να είναι και δικό μα στόχο των Ευρωπαίων και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας στην προετοιμασία ε, της διάσκεψης για τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Αλαφράνκα πρώτο για 1,5 λεπτό από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Και πάλι έχουμε τη Συρία στην ημερησία διάταξη του Κοινοβουλίου. Είναι η 8η χρονιά του πολέμου. Δεν σταματάει η κρίση. Και ε, είναι τρομακτικά τα στοιχεία. Μισό εκατομμύρια ε, νεκροί, 5 ε, εκατομμύρια και οι πρόσφυγε διάφορα παιδιά που ε, υφίστανται τέτοια προβλήματα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια καταστραμμένη χώρα. Είναι πολύ ανησυχητικά αυτά και σε αυτό το πλαίσιο όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. 65% του εδάφους ελέγχει ο Σύρος Πρόεδρος και σύμμαχοι του Ρώση και Ιρανοί. Έχουμε εντάσεις στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ και γενικότερα είναι πολύ ασταθής η περιοχή και αβέβαιη. Και εκεί έχουμε ένα νέο σενάριο ψυχρού πολέμου. Όλοι προς τα εκεί κινούνται. Ε, έστειλαν στο Ισραήλ τον Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας Ηνωμένε Πολιτείε. Οι πρόεδροι Ρωσίας, Ιράν και Τουρκία συνεδριάζουν την Πέμπτη στο Σότσι. Προσπαθεί η Συρία να συνάψει και πάλι συμμαχίες με εταίρους όπως τα Εμμυράτα και η Ορδανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Επίτροπε, τι να κάνει. Είναι πολύ δύσκολο να πάμε πιο πέρα από την κοινή μας ε, στρατηγική, να στηρίζουμε διεθνείς διασκέψεις και να συγκεντρώνουμε κονδύλια που συγκεντρώνουμε. Υποστηρίζουμε τον ειδικό εντεταλμένο και τον οδικό χάρτη των ΗΕ. Αλλά κύριε Επίτροπε, αρκεί αυτό για να ανακουφιστεί ο κόσμος αυτός, η χώρα αυτή, η μαρτυρική Συρία που συνεχίζει να πεθαίνει. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Μποστινάρου, για 1,5 λεπτό επίση. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ορισμένοι λένε ότι ο πόλεμο στη Συρία έχει λήξει. Εγώ νομίζω ότι η δήλωση αυτή δεν είναι σωστή, αποτελεί παρανόηση. Μολονότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση στι εχθροπραξίε, στην πράξη δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδο όσον αφορά τα βαθύτερα αίτια τη σύγκρουση. και η ειρήνη φαντάζει ακόμα τόσο μακριά. Όντως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα στρατεύματα του Ασάντ, του Ιράν και της Ρωσίας έχουν καταφέρει να καταλάβουν επικράτειες που παλιότερα ανήκαν ακόμα και σε τρομοκράτες μαχητές. Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι εξακολουθούν και χρησιμοποιούν απαγορευμένα όπλα. Θα τερματιστεί στην πραγματικότητα ο πόλεμος θα βρούμε έναν τρόπο να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική πολιτική μετάβαση με πραγματική λογοδοσία και πραγματική μεταβατική δικαιοσύνη όταν θα διασφαλίσουμε ότι τα 6 εκατομμύρια των προσφύγων και τα 4 εκατομμύρια των ιστορικά εκτοπισμένων στη Συρία θα έχουν ένα σπίτι στο οποίο να μπορούν να επιστρέψουν και όταν θα μπορεί πραγματικά να του προστατεύει το ίδιο το κράτο του. Τότε θα ξεκινήσει η συγκρότηση, τότε θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση κύριο όρο εδώ πέρα είναι η δικαιοσύνη. Έχουμε πολλά εγκλήματα πολέμου, από συστηματικούς, συστηματικούς βασανιστήρια, από αυθαίρετε κρατήσει, μέχρι την παρεμπόδιση τη ανθρωπιστική βοήθειας και μέχρι τη συστηματική χρήση απαγορευμένων όπλων από το ρουσικό καθεστώ, τη συριακό με καθεστώς και από τις συμμαχικές του δυνάμες. Αν το δικαστικό σύστημα της Συρίας δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει ανεξάρτητες διώξεις και έρευνε, θα πρέπει εμείς να βρούμε μια διεθνή λύση. Και απευθυνόμενο στον κύριο Επίτροπο θα ήθελα να πω το ακόλουθο. Δεν μπορούμε εδώ πέρα εμείς να δεχόμεστα τετελεσμένες καταστάσει που μας προτείνει, μα επιβάλλει ο Μπασάρα Λασάντ και όσοι το προστατεύουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Να Ευχαριστώ εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Κύριε Τάνοκα, έχετε 1,5 λεπτό κι εσείς. Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει επιβιώσει χωρίς καμία αμφιβολία πλέον το καθεστώς του Ασάντ και ουσιαστικά με την αποχώρησή του τα αμερικανικά στρατεύματα μπορεί να αφήσουν ένα τεράστιο κενό ασφαλείας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαχητές όμω του ISIS που παραμένουν σκορπισμένοι στην Συρία και στις ε, γύρω περιοχές και βλέπουμε ότι στην περιοχή του Ιντλίπ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η σύγκρουση αυτή. Χθε ε, συναντήθηκαν ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν περισσότερο την κατάσταση στο Ιντλίμπ και για να δούνε τι μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα με τις αποστρατικοποιημένες ζώνες. 3,5 περίπου χιλιάδε κάτοικοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Ιντλίπ. Θα πρέπει εμεί να ασχοληθούμε λίγο με τι συνθήκε διαβίωσή του, οι οποίε επιδεινώνονται όλο και περισσότερο εξαιτία Τη βίαιης τάσης που κρατά ο Μπασάρα Λασάντ, ο οποίος θέλει να ξανακερδίσει την επαρχία αυτή πάση θυσία. Έχουμε πάρα πολλούς πολέμους αντιπροσώπων, αν θέλετε, που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια της Συρίας και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας απόμακρος παρατηρητής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η δική μας διπλωματική στάση με έναν Μπασάρα Λασάντ, ο οποίο θα παραμένει στην εξουσία. Ευχαριστώ που σου φιλελευθέρωσε, κυρία Σχάκε για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η υπόσχεση να μην επαναληφθούν τα παλαιότερα είναι ε, τελικά βλέπουμε ότι πεθαίνουν στις φυλακές. Ε, αυτό προέκυψε από ένα άρθρο στη Washington Post την περασμένη εβδομάδα για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν ε, στις φυλακές εκεί. Ο Σίζαρ κατάφερε να διαρρεύσει πληροφορίες από εκεί θέτοντας τη ζωή του και αυτή της οικογένειάς του σε κίνδυνο. Η Ευρώπη δεν είναι απλά άλλος ένας παίκτη σε ό,τι αφορά την Συρία. Πρέπει να αλλάξει η σημερινή μας τάση. Ακόμα δεν έχουμε κίνδυνο κοινή ενωσιακή στρατηγική και πρέπει και η αλλαγή πλεύσης στη Συρία έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις ενώ ο ISIS ακόμα δεν έχει νικηθεί. Κατανοώ ότι λέμε ότι μπορεί να υπάρχει μόνο στρατιωτική λύση για τη Συρία, όμω οι στρατιωτικέ κινήσει ε, διαμορφώνουν και το πλαίσιο, την πραγματικότητα επιτόπου. Πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πιέσει, ιδίω σε αφορά την προστασία των ε, αμάχων στο Ιτλίπ και εκεί κοντά. Αλλά και ε, το Χαλέπι και οι Χόμς ε, υπάρχει κίνδυνος να τεθούν στο στόχαστρο και πάλι. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι οτιδήποτε κάνουμε σε ό,τι αφορά τι κυρώσει προ τη Συρία θα υιοθετείται και θα υλοποιείται κιόλα. Έχουμε, για παράδειγμα, κυρώσει και δεν έχει νόημα να επιβάλλουμε κυρώσει αν δεν υλοποιούνται. Αρκεί βέβαια να μην έχει αυτό αντίκτυπο και στον ε, πληθυσμό εκεί. Ακούσαμε ε, ότι οι βελγικέ ε, εταιρείε έχουν αποστείλει τόνου χημικών ουσιών στη Συρία που οδηγούν στην δημιουργία και κατασκευή όπλων και δεν είμαστε τελικά αξιόπιστοι αν δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Τέλος, στο Λίβανο, στην ε, Ιορδανία και στην Τουρκία. Αυξάνεται η πίεση προ ε, τι ε, τοπικέ κοινότητε και οι νέοι και οι πιο ευάλωτε κατηγορίε τίθενται στο στόχαστρο. Πρέπει να αποφύγουμε τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών, αλλά και την δημιουργία άλλων πολιτικών δυνάμεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας κανονικά θα είχε το λόγο, αλλά δεν τον βλέπω από την Αριστερά. Ο κύριος Ραϊμόν από πλευράς Πρασίνων Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ένα μισή λεπτό. Όχι, δύο λεπτά έχετε. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάν, κύριε Επίτροπε, καλώ ορίσατε στην Ολομέλεια. Χαίρομαι που σα βλέπω και θέλω να απευθυνθώ σε εσά ειδικά. Ενώ εμείς συζητούμε εδώ, στη Συρία μπορεί να διεξάγονται οι τελευταίες μάχες με το Ισλαμικό κράτος, από σπίτι σε σπίτι, με Κούρδους και συμμάχους τους, που τις τελευταίες ώρες θα απελευθερώσουν και τις τελευταίες περιοχές. Είναι καταπληκτικό αυτό το επίτευγμα και η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι ευγνώμων γι' αυτό. Αντιθέτω, και πάλι ετοιμαζόμαστε να εγκαταλείψουμε του Κούρδου και του συμμάχου του. Η αυτόνομη περιφέρεια στη βόρεια Ανατολική Συρία είναι και δημοκρατική και πολυπολιτιστική. Είναι γεζιντή και χριστιανοί, δεν είναι μόνο Κούρδοι και πολλοί Άραβε, ε, λαϊκοί, κοσμικοί και εκεί είναι περισσότεροι πλέον μαχητέ, άνδρες και γυναίκε, άραβε παρά Κούρδοι. Προσπαθούν δημοκρατικά να στήσουν μια αυτόνομη περιφέρεια και έχουν προχωρήσει πολύ. Και έχουν και σχολιά, έχουν και νοσοκομεία, επενδύουν με μικρή υποστήριξη από την Ευρώπη. Και τώρα ε, τους απειλεί τουρκική εισβολή με τον Ερτογάν ο οποίο θέλει να περάσει τα σύνορα και να εισφάλει στην περιοχή αυτή. Και η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για να του προστατεύσει. Εσεί που είστε και επίτροπο γειτονία παρακαλώ ασκήστε μεγάλη πίεση στην Τουρκία. Εάν συμβεί αυτό το σχέδιο της ε, Τουρκίας ε, και καταστρέψει τη βορειοτολική Συρία, πρόβλημα έχει και η Ευρώπη. Υπάρχουν εκεί στις φυλακές 900 Ευρωπαίοι πολίτες μαχητές του ISIS και τους φυλάνε οι Κούρδοι και είπανε ότι δεν θα τους σκοτώσουμε, αν μπει ο Ερντογάν θα τους αφήσουμε ελεύθερους και θα έχουμε 900 μαχητές, τρομοκράτες, αδέσποτους που θα πάνε στην Ευρώπη. Ε, έχουμε πολύ μεγάλο συμφέρον να μην γίνει εισβολή, να υπάρχει ειρήνη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να είμαστε στο πλευρό των Κούρδων συμμάχων τους και των δικών τους συμμάχων και να είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστώ. Από την ομάδα EFTT ο κύριος Κάρβερ για 1,5 λεπτό. Επίτροπε, το ε, μήνυμα που μπορώ να ε, μεταφέρω από την επίσκεψη τον Δεκεμβρίο είναι ότι τελικά όλα αυτά έχουν ε, φέρει κοντά τις προηγουμένως αντιθέμενες δυνάμεις ενώπιον του κοινού εχθρού. Υπάρχουν επιφυλάξει ό,τι αφορά και τι πρόσφατε διακηρύξει του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσουν οι Αμερικανικέ δυνάμει από τη Συρία. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ελαττώματα στην προσέγγιση μα, όμω δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την δημιουργία κενού που μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι θέλουν να προωθήσουν τη δική του ατζέντα. Ε, οι Κούρδοι, για παράδειγμα, θα πρέπει να ε, παραμείνουν ε, και να διατηρηθεί η ισορροπία στην περιοχή σε σχέση και με τι διάφορε ομάδε που υπάρχουν στι κοινωνίε τη Μέση Ανατολή. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν του σαφεί κινδύνου, αλλά να θυμόμαστε ότι χωρί τη Δύση και χωρί την Αμερική τελικά τι απομένει. Πρέπει ρεαλιστικά να αναγνωρίσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Αν δεν επηρεάζουμε εμεί, θα επηρεάσουν άλλοι την περιοχή και δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε καμία περίπτωση το πιθανό ε, αποτέλεσμα. Πρέπει να προσεγγίσουμε το μέλλον τη Συρία και για την μελλοντική ευημερία του ε, Συριακού λαού, αλλά και για την δική μα ε, ασφάλεια και επιρροή στη Δύση με έναν σόφρονα τρόπο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη ομάδα ΕΝΕΦ, κυρία Αγνοτού, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι ατλαντιστικές δυνάμεις καθώς επίσης και οι δικτατορίες που βασίζονται στα πετροδολάρια οι οποίες υποστήριξαν και ουσιαστικά εξόπλισαν τους Ισλαμιστές, δεν είναι πλέον οι κύριοι του παιχνιδιού στη Συρία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Από την άλλη υπάρχει μία δαμόκλειο σπάθη πάνω από τις κυβερνήσεις μας και πάνω από τους πολίτες μας. 450 Κρατούμενου έχουμε αυτή τη στιγμή, ριζοσπαστικοποιημένου. 50 τζιχαντιστέ οι οποίοι θα απελευθερωθούν σύμφωνα με την κυρία Νικόλ Μπελουμπέ, η οποία είναι υπουργό δικαιοσύνη τη Γαλλία. Ο κύριο Κριστόφ Καστανέρη, υπουργό Εσωτερικών, είπε ότι θα επιστρέψουν στη Γαλλία ακόμα 130 μαχητέ. Στο Βέλγιο είδαμε ότι απελευθερώθηκαν 182 Ισλαμιστέ από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρή νομοθεσία, θα πρέπει να είναι απόλυτη η αυστηρότητά μα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αφαιρέσουμε την υπηκότητα από όσου Ισλαμιστέ έχουν διπλή υπηκότητα. Όσον αφορά του εξτρεμιστέ που ζουν στη δική μα τη χώρα με μία μόνο εθνικότητα, ε, για αυτού θα πρέπει να προβλεφθούν τα κάτεργα ή ακόμα και θαντική ποινή. Πρόκειται για προδότε και ω τέτοιοι θα πρέπει να τιμωρηθούν. Μία διαγραμμένο τώρα, το λόγο έχει ο κύριο Ζαριανόπουλο. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποχωρούν ουσιαστικά από τη Συρία. Αναδιατάσσουν τι δυνάμει του στην περιοχή, αναβαθμίζουν την παρουσία του με το ιράν πάντα στο στόχαστρο μέσα σε ένα κουβάρι οξύδα των αντιθέσεων με το δάχτυλο στη σκανδάλη και ταυτόχρονα παζάρια με ρωσία ισραήλ χώρε του κόλπου την αίγυπτο. την τουρκία βεβαίω σε αναβαθμισμένο ρόλο που επεμβαίνει ανενόχλητη στρατιωτικά στην περιοχή. σχεδιάζεται ο μεταπολεμικό έλεγχο ολόκληρη τη μέση ανατολή και τη νοτιοανατολική μεσογείου. στην ίδια βέβαια κατεύθυνση η ευρωπαϊκή ένωση η γαλλία η βρετανία η γερμανία η ιταλία επεμβαίνουν στρατιωτικά και επιχειρηματικά πατρονάρουν τριμερείς άξονες όπως ισραήλ κύπρο Ελλάδα, με την τελευταία υποκυβέρνηση σύριζα σε ρόλο μεντεσέ και σημεοφόρου διάβλου επικοινωνία του με την τουρκία όταν δυσκολεύουν τα παζάρια. μεταξύ άλλων μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο η κύπρος με μεθόδευση διχοτόμησής τη υπονατοϊκή ομπρέλα πέραν βεβαίως των τουρκικών διεκδικήσεων κατά της ελλάδας. Καταραίει ο μύθο λοιπόν τη κυβέρνηση σύριζα ότι οι ηνωμένες πολιτείες νάτο και ευρωπαϊκή ένωση διασφαλίζουν ειρήνη στην περιοχή. μόνο ανταγωνισμού, πόλεμο και δυστυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ ε, από τι πολιτικέ ομάδε. Ακολουθούν τώρα οι λοιποί ομιλητέ. Ο κύριο Τόκε, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Συρία σοβεί ένας φωνικός πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα τη μοίρα των χριστιανών που διώκονται. Σύμφωνα με μια μελέτη της Open Doors, 70 χώρες είναι εκείνες που διώκουν χριστιανούς. Ο χριστιανισμός είναι από τις πιο διωκόμενες θρησκείες παγκοσμίω. Στη Συρία βλέπουμε η χώρα να βρίσκεται στην ενδέκατη θέση αυτού του θλιβερού καταλόγου και έχασε τους μισούς χριστιανούς κατοίκους της κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι θετικό αυτό, έχει δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Ε, φυσικά αυτό δεν φτάνει απέναντι σε αυτή τη μόνιμη και διαρκή κρίση. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αίτια του πολέμου. Ο πόλεμος στη Συρία θα πρέπει επιτέλους να τέρματιστεί. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για τους πρόσφυγες ε, θα πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα το ουγγρικό μοντέλο. Δηλαδή η καλύτερη εναλλακτική στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι απλώ να υποδεχόμαστε εκατοντάδε χιλιάδε προσφύγων, αλλά να εξασφαλίζουμε την ασφαλή επαναπατρισμό του. Ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να εισάγουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη, αλλά να δίνουμε βοήθεια επιτόπου για να λύνονται εκεί. Στην Ουγγαρία, γι' αυτό το λόγο, ε, δημιουργείται ε, γραμματεία σε ένα Υπουργείο ε, που ασχολείται, Γενική Γραμματεία, με την επιστροφή των χριστιανών και την ανοικοδόμηση της Συρίας. Άρα, εκεί θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές. Η κυρία Βαλενθιάνο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά, ε, νομίζετε ότι ανήκει στο παρελθόν ο πόλεμος στη Συρία Είδαμε εδώ να φτάνουν ε, ποτάμια προσφύγων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τη φρίκη. Φυσικά και είναι ανοιχτό το μέτωπο. Ήταν πολύ μεγάλες οι αυταπάτες. Ε, έχουμε τον παλιό ψυχρό πόλεμο και τον καινούργιο ψυχρό πόλεμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Κίνα ε, συστηματικά ακύρωναν οποιαδήποτε συμφωνία. Όπως και πάντα η Ευρώπη έχει τύψεις και προσπαθεί να βοηθήσει ε, τον λαό της Συρίας μετά από αυτή την έξοδο. Αλλά μετά από 10 χρόνια φρίκης έχουμε αρχαίες πόλεις ε, ε και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ε, στις ρώσικες ε, βόμβες ή στα ντρόνς των ΗΠΑ έπεσαν θύματα. Και τώρα τι θα γίνει. Αυτό δεν μπορεί να τερματιστεί χωρίς να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι υπέτειοι. Ο πόλεμος σταμάτησε ε, την τυραννία του Ασάντ, αλλά πού είναι η δημοκρατική αντιπολίτευση. Ποιο τη θυμάται, κανεί. Και τώρα κινδυνεύουν ακόμα και οι Κούρδοι. Η τρίτη διάσκεψη για το μέλλον τη Συρία έρχεται την ώρα που θα πρέπει να συζητήσουμε για ευθύνε. Θα συζητήσουμε για το μέλλον χωρίς ε, να σκεφτούμε ότι υπάρχει καταστροφή, λες και δεν έγινε. Αυτό θα πρέπει να ζητήσει το Κοινοβούλιο. Ευθύνε. Δεν θα πρέπει να, να περάσει αυτή, αυτή η κατάσταση και αυτή η φρίκη. Ο κύριος Μπέλντερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική που ακολουθείται από την ε, Τουρκία δεν μπορεί να μας αφήσει ε, ε, ήσυχους. Πρέπει να δούμε την προσέγγιση που ακολουθεί δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις το 2016 και το 2018 έχουν μετατρέψει ε, σε προτεκτοράτο ε, της Τουρκίας δύο περιοχές ε, της Συρίας και θέλουν να δημιουργήσουν μια τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Συρίας όπως έγινε και με την Κύπρο. Οι τουρκικές διακηρύξεις σε ό,τι αφορά την εδαφική ακαιρεότητα φαίνεται ότι είναι μόνο λόγια. Ε, μιλούν βέβαια και για τον κουρδικό κίνδυνο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ε, θέλουν ουσιαστικά να καθαρίσουν ε, τις χριστιανικές περιοχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα ενωσιακά συμφέροντα, αλλά πρέπει να μας μιλήσετε περισσότερο και για τον ρόλο της Τουρκίας. Το αναφέρατε, αλλά πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάουτμαντ για το λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολλοί συνάδελφοι ήδη το ανέφεραν. Εδώ και 8 χρόνια ε, διαρκεί αυτός ε, ο πόλεμος ε, στην Συρία. Κάτι που ξεκίνησε ως ειρηνική, ειρηνικές διαδηλώσεις για τη δημοκρατία, τελικά οδήγησε σε πραγματική αιματοχυσία. Σε όλη την χώρα έχουμε πάρα πολλά θύματα πάνω από 465.000 Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή του, 1 εκατομμύριο τραυματισμένοι και 12 εκατομμύρια, σχεδόν το ίμιση του πληθυσμού, αναγκάστηκε να φύγει. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η κατάσταση και σήμερα ε, και το Ισραήλ ε, ε, παρέχει τα όπλα και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το δικό τους ρόλο Έχουμε και τους Κούρδους ε, που ε, πλήττονται από τουρκικούς βομβαρδισμούς και επιπρόσθετα έρχεται και ο Τραμπ να μας πει ότι αποσύρει ε, τα στρατεύματά του επειδή ο ISIS έχει νικηθεί, παρότι οι δικοί μας λένε το κάτι διαφορετικό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σήμερα εδώ στο ημικύκλιο, βλέπουμε ότι μιλούμε για μία από τις πιο αιματηρές σειράξεις, όπου ε, ε, έχουμε βομβαρδισμούς αμάχων, ε, γυναικόπαιδα ζουν σε καταβλισμούς εδώ και 8 χρόνια και τελικά τίποτα δεν γίνεται. δεν υπάρχει ψυχή, όπως και εδώ σήμερα, όταν συζητούμε τέτοια θέματα. Ελπίζω μόνο στην Ευρώπη και εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε κάτι διαφορετικό επιτέλους. Να υπάρξουν πραγματικά κυρώσεις, να πιάσουμε την πραγματική αιτία του προβλήματος εσείς και εγώ κύριε Επίτροπε έχουμε γεννηθεί σε μια ειρηνική χώρα, σε μια χώρα που διάγει περίοδο ειρήνης. Ε, δεν μπορώ να πούν το ίδιο δυστυχώ ε, τα παιδιά που γεννιούνται εκεί στην Συρία. Αν είχα τι λύσει, θα σα τι έλεγα βέβαια. Εσεί όμω είστε καλύτερο και πιο σοφό. Πρέπει λοιπόν να κάνετε ό,τι μπορείτε για να ε, βάλουμε ένα τέλο σε αυτή τη ε, διαμάχη. Ευχαριστώ. Κύριε Ορμπάν Κρέσπο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Συρία είναι κατάφορο παράδειγμα αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας, αλλά ακόμα ένα παράδειγμα της υποκρισίας της. Ποιος κέρδισε το Ισλαμικό κράτος, οι Κουρδοί, ο κουρδικός λαός. Και τώρα τους εγκαταλείπουμε στη μοίρα τους, απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν και Τουρκίας. Από εδώ εμείς κάνουμε τα στραβά μάτια όταν επιτίθενται στον άμαχο πληθυσμό και ε, τους λαιλατούν, τους παίρνουν τις πηγές όπως είναι οι ε, τόνοι ε, από ελιές που έρχονται από το Αφρίν και φτάνουν στην Ευρώπη, στην Ισπανία εμπροκειμένα. Η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί στο πολιτικό διάλογο, στο διεθνή διάλογο, στην ε, προώθηση του διεθνούς δικαίου για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Θα πρέπει ο κουρδικός λαός να εξασφαλίσει τα κοινωνικά και πολιτικά του επιτεύγματα, όπως είναι η ισότητα του φύλου. Να μην τους βήσουν από το χάρτη τώρα που ε, απειλεί να εισβάλλει στις τουρκικές περιοχές ο τουρκικός στρατός. Και στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κόψει τις προτιμησιακές συμφωνίες συμφωνίε με την Τουρκία που λέει λατή το κουρδικό ε, ε, λαό και εκτό τη Τουρκία. Όλα τα άλλα είναι ωραία λόγια και ψηφίσματα που κρύβονται κάτω από γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που δεν ανταποκρίνονται στα συμφέροντα ε, ούτε τη Συρίας ούτε τη πλειονότητα του κουρδικού λαού. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ορμπάν Κρέσπο. Η κυρία Σόιτροβα έχει γαλάζια κάρτα. Συμφωνείτε, δέχεστε μια μπλε κάρτα ερώτηση. Παρακαλώ, κυρία Σόιτροβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ σας κύριε συνάδελφε που δέχεστε την μπλε κάρτα. Συμφωνώ ότι η Τουρκία και ο Ερντοάν ε, καταχράται εκεί και εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να επιτεθεί στους Κούρδους. Ε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πραγματικά την κατάσταση που επικρατεί εκεί για να περιορίσει και να καταπιέσει τις, τουρκικές, τις κουρδικές συγγνώμη, μειονότητες. Πάντως διαφωνώ μαζί σας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. Τι ευθύνη έχει η διεθνής κοινότητα για ένα εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2013 στη χώρα. Ο κύριος ε, Μπαρόν Ουρμπαν ε, Πολλές ερωτήσεις ε, κάνατε. Εγώ μίλησα για την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννοούσα τις προτιμησιακές συμφωνίες που έχουμε με την Τουρκία. Δεύτερον, επιτρέπουμε να έρχονται ελιές από το Αφρίν, ε, τις κλέβουν από τον κουρδικό λαό και τις πουλάει η τουρκική κυβέρνηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή είναι η ευθύνη και έχει ευθύνη και η διεθνή κοινότητα και τα διάφορα συμφέροντα ε, που έχουν μπει στον πόλεμο στην Τουρκία και είναι ε, Τελείω ξένα προς το Συριακό ή τον Κουρδικό λαό. Αυτά εννοούσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάσταση στη Βόρεια Συρία παραμένει απειλητική. Από τη μια η Τουρκία επανειλημμένα έχει απειλήσει ότι θα επέμβει στρατιωτικά κατά των κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή Ρατζάβα. Ταυτόχρονα η ε, Συριακή κυβέρνηση ανακτά εδάφη και το Ιτλίπ όπου περίπου 3 εκατομμύρια άμαχοι ζουν και πολλές ένοπλες ε, ομάδες σοβούν η ε, στρατιωτική ε, προώθηση της Τουρκίας ή της Συρίας ε, στη Βόρεια Συρία θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθούν. Η ευρωπαϊκή διπλωματία να εξακολουθεί να πιέζει για την επανάληψη συνευτικών συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και ΠΚΚ. Στη διάσκεψη των Βρυξελών για τους δωρητές θα πρέπει να είναι ισομερός και κατάλληλα εκπροσωπημένη και η γνώμη και η κοινωνία των Υπάρχουν και μεγάλα προγράμματα επαναπατρισμού ε, και μετεγκατάστασης και θα πρέπει να υπάρχουν και ασφαλείς οδοί στην Ευρώπη. Κύριο κύριος Μάρουζικ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν η Συρία βρισκόταν σε άλλο σημείο του πλανήτη, κανείς δεν ενδιαφερόταν για τη χώρα αυτή. Ήθος ε, λοιπόν να μην έχουμε εκεί τη χειρότερη κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και χειρότερε χώρε και χειρότερε κυβερνήσει. Αυτό όμω δεν είναι τόσο πρόβλημα τη Συρία, όσο γενικότερο ζήτημα τη ε, Μέση Ανατολή. Γιατί στην περιοχή αυτή έχουμε επιθέσεις και εχθροπραξίες από διάφορες δυνάμεις και από διάφορες χώρες. Έχουμε το Ιράκ, την Λιβύη, την Αίγυπτο, παράγοντες, χώρες μάλλον οι οποίες καταστράφηκαν στο παρελθόν εντελώς, χώρες στις οποίες εκτελήθηκαν τεράστια ανθρώπινα δράματα και για τις οποίες δεν μιλάμε ποτέ. Επικεντρώμαστε μόνο στη Συρία. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, ποια είναι τα βαθύτερα αίτια από όλες αυτές τις συγκρόσεις, θα πρέπει να ζητήσουμε την αλήθεια, τα πραγματικά αίτια της εξωτερικής στρατιωτικής παρέμβασης σε διάφορες περιοχές. Ποιος πουλεμά και για ποιο λόγο, ποιος καταστρέφει εκ από έξω τις χώρες αυτές. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση ορθολογικά να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Κύριε Πιτίδη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά την ε, ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον ε, πρόεδρο Τραμπ περί της αποχωρήσεως των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία ε, η κατάσταση στη μέση ανατολή έχει μεταβληθεί έχει γίνει περισσότερο συγκεκριμένη. η απόφαση για την αποχώρηση ελήφθη χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους ε, υπολείπους εμπλεκομένους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα κενό το οποίο όλοι προσπαθούν να καλύψουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Στον ελάχιστο χρόνο που μου διατίθεται δεν μπορώ να κάνω μια σε βάθος ανάλυση της καταστάσεως. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι ενώ στη σκακέρα της Συρίας όλοι οι παίκτες ε, κερδίζουν πλεονεκτήματα η μόνη απούσα είναι η ευρωπαϊκή ένωση έχοντας επιλέξει να είναι από την αρχή της κρίσεως και του πολέμου η ουρά της πολιτικής των ηνωμένων πολιτειών τη στιγμή αυτή αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα. ο ένας είναι από την αναβαθμισμένη τουρκία. αντιλαμβάνεστε ότι η επιθετικότητα και η προκλητικότητα της τουρκίας τώρα θα αυξηθούν ο δεύτερο κίνδυνο είναι από του ε, φανατικού τζιχαντιστέ του isis οι οποίοι αν και ιτήθηκαν στρατιωτικά έχουν διασωθεί και ετοιμάζονται να επιστρέψουν με διαφόρου τρόπου στι πατρίδε του στην ευρώπη για να αναλάβουν τρομοκρατική δραστηριότητα. ευχαριστώ. Κύριε Επίτηδε, κύριε Επίτηδε, με ακούτε σας παρακαλώ κύριε Επιτίδιε. Έχετε μπλε κάρτα. Ε, συμφωνείτε, παρακαλώ, από τον κύριο Έθριτζ. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτηση. Θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι το παράδειγμα της Συρίας είναι πολύ το παράδειγμα ότι όταν κάποιος αρχίζει να βομβαρδίζει από το εξωτερικό και να επεμβαίνει στρατιωτικά ε, ε, λένε ότι υποστηρίζουν τη δημοκρατία και μετά έρχονται οι Ρώσοι και επιτίθενται στο ISIS και τα λοιπά, αλλά έτσι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και τα προβλήματα. Και τουλάχιστον ο κύριος Τραμπ ε, προτείνει να φύγει και να αφήσει τον κόσμο να ζήσει τη ζωή του μόνος του εκεί. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτησή σας. Ε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο απλά λέω αυτό. Έτσι ακριβώς όπως παρουσιάσατε τα πράγματα, αυτό δυστυχώς συμβαίνει και αυτό δεν βοηθά την ε, γενικότερη πολιτική, την αξιοπιστία, αλλά και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μεγιάν Μόν. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πόλεμος στη Συρία είναι πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Δεν μπορεί κανείς να το συζητήσει ε, σε λίγα λεπτά. Έχει πολλές πλευρές, ε, πολλά εμπλεκόμενα μέρη και βαθιά εμπλεγμένα τρίτα κράτη. Εδώ με ανησυχεί η μικρή επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο γιατί ανήκειλαν υποχώρηση ε, στρατευμάτων. Και επίση το καθεστώ στη Δαμασκό, εκτό από αυτού, αποφασίζουν και το Ιράν και η Ρωσία και η Τουρκία. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ε, επιρροή. Ε, δεν πρόκειται μόνο για την ήττα του Νταέσε και αυτού του Ισλαμικού κράτους. Πρέπει να αρχίσει μια πολιτική διαδικασία και να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας η πλειονότητα του λαού. Η χώρα είναι μεσογειακή πολύ κοντινή. Ό,τι συμβαίνει εκεί έχει επιπτώσεις και σε εμά. Και σκεφτείτε τη μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 και τις τεράστιες ε, πιέσεις που γνωρίσαμε στα σύνορά μας. Θα πρέπει εμείς να επηρεάζουμε περισσότερο και το παρόν και το μέλλον στη Συρία. Και τέλος, Επίτροπε, θα ήθελα να μας πείτε εάν υπήρξαν αποτελέσματα από την πρόσφατη συνάντηση της κυρίας Μογκερίνη με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν από λίγες μέρες, ε, ο πρώην υπατός εκπρόσωπος της Ένωσης, Χαβιέρ Σολάνα, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο ε, από τον Άσαλτ στον Άσαλτ μέσω κολάσεως. Αυτό είναι λοιπόν η απόλυτη ε, αποτυχία σε ένα πόλεμο χωρίς κανένα νόημα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι κατέστρεψαν το μέλλον τους. Δεν έχει σβήσει η φωτιά αυτή τη κόλαση, αλλά έχει έρθει η στιγμή να σκεφτούμε την ανοικοδόμηση, την ηλική ανοικοδόμηση προφανώ, αλλά κυρίω την ανοικοδόμηση τη ζωή εκεί των πιο νέων. Τα παιδιά αυτά, που είναι εκατομμύρια παιδιά, που έχουν χάσει τα σχολιά του, που έχουν χάσει το ίδιο του το μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευθεί ε, σε ένα πολιετές σχέδιο για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Όχι μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και με συνεργασία αναπτυξιακή. Αυτό είναι ο βασικός στόχος που θα πρέπει εμείς να προωθήσουμε στην τρίτη διάσκεψη ελεγγύης με τη ΣΥΡΙ. Ε, Κύριε Βίστησεν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τραγική η κατάσταση ε, ε, και αυτά που συμβαίνουν. Ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει εξωτερική πολιτική. Καταδικάσαμε τους Αμερικανούς γιατί επενέβησαν και τώρα έχουμε στην πίσω αυλή μας ένα χάος. Η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν ανακατεύονται εκεί και έχουν και συμφέροντα η Ευρώπη τι κάνει. Ποιος κέρδισε. Οι Κούρδοι που αγωνίστηκαν κατά του Ασάτ και του Ισλαμικού κράτους που ήταν οι δικοί μας σύμμαχοι ε, θα την πληρώσουν τώρα. Ποια είναι η λογική συνέπεια. Η κριτική ε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη δεν είναι καινούρια. Είναι από την εποχή του Αφγανιστάν και του Ιράκ οι Αμερικανοί ε, αρνούνται να λύσουν τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Ε, αυτή είναι η πολιτική τους, αλλά η διατλαντική ε, συνεργασία και σχέση είναι ένα ασφαλιστικό δίκτυο για την Ευρώπη. Είναι αντιπαραγωγικό να κατηγορούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Σόιδροβα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δίδεται η ε, επιφανειακή εντύπωση ότι η η κατάσταση στη Συρία, αλλά στην πραγματικότητα η χώρα είναι εντελώ κατεστραμμένη. Το καθεστώ του Ασάντ έχει κερδίσει τον πόλεμο χωρί να έχει την νομοποιήσει όμω από το λαό του. Το καθεστώ του Ασάντ παραμένει με τη βία στην εξουσία με τη βοήθεια τη Ρωσία και του Ιράν. Εκατοντάδε χιλιάδε οι πρόσφυγε από τη Συρία δεν ξέρουν πού να πάνε και αναγκάζονται πολλέ φορέ να επιστρέψουν, μολονότι κινδυνεύουν με δίωξη και με καταδίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε οποιαδήποτε επίθεση της Τουρκία, στο Ιντλίπ γιατί θα έχουμε μία ακόμα ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτό που μας ανησυχεί όμως ακόμα περισσότερο είναι η επιρροή του ίδιου του Ιράν το οποίο φέρνει σε αντιπαράθεση όλο και περισσότερο τη χώρα αυτή με το Ισραήλ. Κάποιες πληροφορίες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες Μα καταδεικνύουν όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει εξωτερικό παρατηρητή, ενώ οι Κούρδοι τελικά είναι οι μόνοι οι οποίοι δίνουν πραγματική μάχη με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει σημαντικότερε διπλωματικέ προσπάθειε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τι προοπτικέ των παιδιών εκείνων που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, που είναι πραγματικοί όμοιροι του Ασάντ. Κύριε Μπενιφέ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Συρία απέχει πάρα πολύ από τον λυθεί και σε μερικέ εβδομάδε έχουμε την τρίτη αυτή διάσκεψη για τη Συρία που διοργανώνει η ύπατη εκπρόσωπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τη δικασία τη Γενέβη για την ειρήνη βάσει του ψηφίσματο 2254 του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και να υπάρχουν συγκεκριμένε ποινικέ πλέον ευθύνε για του εγκληματίε πολέμου. Παράλληλα όμω η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει περισσότερο ω ανθρωπιστικό παράγοντα. Θα πρέπει να βοηθήσει κατά τρόπο ανθρωπιστικό τον Συριακό λαό που δεν το έχει κάνει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να προσκληθεί και στην τρίτη αυτή διάσκεψη. Α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσει όπω η Κολόμπα, η οποία έχει δημιουργήσει ανθρωπιστικού διαδρόμου προκειμένου να βοηθήσουμε του αποκλεισμένου πληθυσμού τη Ρησία. Τα παραδείγματα αυτά θα πρέπει να τα ακολουθήσουν και άλλε κυβερνήσει και άλλοι οργανισμοί. Ο Ιερέα Παύλο Νταλόλιο είχε πει στο παρελθόν στα πλαίσια του διαθρησκευτικού διαλόγου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθούμε όλο και περισσότερο τον διάλογο αυτό. Α καταφέρουμε να προωθήσουμε στον τόπο περισσότερο τα διδάγματα του ανθρώπου αυτού και α δώσουμε όλη μια μάχη για την απελευθέρωσή του. Ο κύριος Ντροτζεύσκη, η κατάσταση στην Συρία δεν έχει επιληθεί. Και αυτό αποδεικνύεται και στην σημερινή συζήτηση από το μεγάλο αριθμό διαφορετικών αναλύσεων της κατάστασης. Να σας πω ένα όμως σημαντικό ε, σκέλος ε, της υπόθεσης. Για όσους ε, από εσάς εξετάζουν το θέμα της Συρίας από οποιαδήποτε προσέγγιση, δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτα. Δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, δεν υπάρχει καμία ανάληψη δράσης Ιδίω του τελευταίους μήνε. Και δεν υπάρχουν συνέπειες σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τα θέματα πρέπει να επιληθούν. Και στρέφω την προσοχή σα σε αυτό, γιατί αυτό είναι και ο λόγο που δεν σημειώνουμε επιτυχίε. Ξέρουμε ότι πιο σημαντικοί φορεί εκεί, η παίκτε, είναι η Ρωσία, η Τουρκία και ο Ασάντ. Στι σημερινέ συνθήκε, σε αυτό το κουβάρι που έχει δημιουργηθεί, αυτοί έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώ δεν είναι καλά για την χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκίλ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, χθες υπήρξε η επίθεση προς ε, τις ε, τελευταίες ε, περιοχές που ελέγχει ο ISIS. Οι τοπικές κοινότητες έχουν συμφωνήσει να δημιουργηθεί ένας διάβλος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες βλέπουμε ότι δεν επαρκούν. Πρέπει να αυξηθούν οι υπηρεσίες περίθαλψης, το νερό και η τροφή. Είναι θετικό λοιπόν και που δημιουργείται και διοργανώνεται αυτή η επίκαιρη ε, εκδήλωση τον ε, Μάρτιο για την περιοχή. Όμω, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η συνδιάσκεψη αυτή δεν θα επικεντρωθεί μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά θα κινητοποιήσει ε, διεθνή και περιφερειακή στήριξη προ την εξέβρεση μια πολιτική λύση. Δεύτερον, η πολιτική μετάβαση πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για, για οποιαδήποτε νέα ενωσιακή επένδυση η απόφαση Τραμπ απόσυρση των δυνάμεων από την Συρία βλέπουμε ότι έχουν οδηγήσει ε, τον ε, Συριακό Δημοκρατικό Στρατό ε, να ακολουθήσει νέα προσέγγιση. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος τελικά στη δυνατότητα στήριξης μιας πολιτικής μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Γκίλ. Κυρία Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει μπλε κάρτα για σας. Συμφωνείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Ναι, παρακαλώ κύριε Ζεμπόρσκα. Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο παρεξήγηση. Ζητούσε το λόγο για το Κατσιάη, κυρία Ζαμπόρσκα, όχι για την μπλε κάρτα. Ζητώ συγγνώμη. Ο κύριο Δία Δεμέρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο πόλεμο στην Συρία έχει δημιουργήσει 6,3 εκατομμύρια πρόσφυγες, 6 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπιστέντες και περίπου 500.000 νεκρούς είναι τραγωδία, η μεγαλύτερη στην πρόσφατη εποχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι, αλλά όχι μόνη τη. Και καλό είναι που το Μάρτιο έχουμε την τρίτη διάσκεψη Ένωση και Ηνωμένων Εθνών για το μέλλον τη Συρία και τη περιοχή. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να συλλέγουμε ανθρωπιστική βοήθεια πάνω από το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με πολιτική πλαισίωση για να καταλήξουμε σε διαπραγματεύσει και ειρηνική λύση. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει ο ΙΕ το ψήφισμα 2254 να εφαρμοστεί γίνεται λόγος για οριστική ήττα ε, ούτε οριστική θα είναι ούτε ήττα ούτε τέλος πολέμου. Ε, χρειάζεται η Συρία τη διεθνή κοινότητα αλλά με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Είναι απαραίτητη η ασφαλής επιστροφή. Ε, είδαμε τους εργά που έχουν έρθει και εδώ στο κοινοβούλιο και τους χειροκροτήσαμε. Ε, ολόψυχα έχουν και τη συμπάθειά μας και την υποστήριξή μας, όλων μας. κοιτάξτε, για να καταλάβουμε όταν ζητάτε το λόγο για το Catch the Eye, μη μου σηκώνετε την μπλε κάρτα, αλλά ένα λευκό χαρτί ή το χέρι σας. Γιατί αλλιώς νομίζουμε ότι ζητάτε να κάνετε ερώτηση στον ομιλητή. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένε ε, ζώνε απαγόρευση των πτήσεων προκειμένου να προστατευθεί ο λαό τη Συρία. Αλλά στην πραγματικότητα δεν προστατεύεται τη στιγμή που το καθεστώ Ασάντ εξακολουθεί και υφίσταται. Τα αποτελέσματα θα έλεγα ότι είναι πραγματικά καταστροφικά στην Συρία όσον αφορά την εξοπιστία και το κύρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φαίνεται σε μια πρόσφατη έρευνα, όπου φαίνεται ότι η εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώ επιδεινωμένη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει αφόρητα στην Συρία, άνθρωποι που έχουν δώσει ολόκληρη μάχη για να αντιμετωπίσουν τρομοκράτες. Κατεφημισμό τους αποκαλούμε ξένους μαχητές. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς είναι Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι που στρατολογούνται και κατατάγονται στα τάγματα του Νταέσ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ε, είναι οι Κούρδοι αυτοί, σύμμαχοι των Αμερικάνων, οι οποίοι δίνουν τη σημαντικότερη μάχη κατά των τρομοκρατών αυτών. Η δική μας υποστήριξη δυστυχώς θα πρέπει να μάλλον δεν πρόκειται να διαρκέσει όσο θα περιμένουμε. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει πέρα από τη διπλωματική υποστήριξη να καταφέρουμε να παράσουμε και την απαραίτητη ανθρωπιστική υποστήριξη. για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχω μεταβεί δύο φορές στη Σύρια. Συνάντησα εκεί ε, εκπροσώπους ε, της χριστιανικής μειονότητας στο Χαλέπι, στη Χόμς και στη Δαμασκό. Κατάλαβα ξεκάθαρα ότι οι κυρώσεις και οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς κατά του συριακού καθεστώτος πλήττουν εκατομμύρια πολιτών, απλών σύρων πολιτών που είναι άνεργοι, χωρίς εισόδημα και αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα τους. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους ανθρώπους αυτούς για να παραμένουν στην πατρίδα τους. Η Ουγγρική κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες αποφάσισε να υποστηρίξει το σύστημα υγείας ε, με το σύστημα ανοιχτά νοσοκομεία στο Χαλέπι και στο Χόμς, ε, ανεξαρτήτως θρησκείας και προέλευσης. 3.640.000 άνθρωποι ε, είναι ε, στην Τουρκία έτοιμοι να φύγουν. Να φύγουν από την Τουρκία, αλλά να μην έρθουν στην Ευρώπη, να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ευχαριστώ ο κύριος Φρόιντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα μεγάλο ερωτηματικό ε, ίσως ερωτηματικό, ελπίζουμε, θαυμαστικό να τελειώνει ο πόλεμος. Έχουμε ζήσει τις επιπτώσεις. Φυσικά, Ποιο, είναι, τι είναι το δικό μας υποτιθέμενο προσφυγικό δράμα απέναντι σε αυτά που έχουν ζήσει οι ε, Σύροι. Έχουν αφήσει τα σπίτια τους για να πάνε να βρουν σε γειτονικά κράτη ε, σωτηρία. Ε, όταν γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο. Θέλω και πάλι να απευθύνω μια έκκληση. Στο μέλλον δεν επιτρέπεται να παραμένουμε απαθείς θύετές αν ξεσπάσει και άλλη σύραξη. Η ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια κοινή εξωτερική πολιτική ισχυρή με διπλωματική παρέμβαση, ε, με αυτοπεποίθηση ε, ως διαμεσολαβητές και εγκαίρως. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποστούμε από την ομοφωνία. Για τη Συρία είναι δυστυχώς πολύ αργά, αλλά πολύ φοβούμαι ότι η Συρία δεν θα είναι η τελευταία χώρα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εξοπλισμένοι εμείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει ε, μπλε κάρτα. Συμφωνείτε να απαντήσετε στον κύριο Ρούμπιχ. Βεβαίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φρόιντ ε, που έθεσε αυτό το κομβικό ζήτημα και ερώτημα. Ε, τη ασφάλεια των ε, σύρων πολιτών. Έχω πάει στον Καζιαντέπ εγώ, στον προσφυγικό ταυλισμό με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και οι περισσότεροι πρόσφυγες στην πατρίδα τους θέλουν να γυρίσουν. Είναι εκεί με τα αυτοκίνητά τους και περιμένουν να τους δοθεί το πράσινο φως για να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καμιά πιθανότητα στο τέλος, ε, ε, στο μέλλον, να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη αποστρατητικοποιημένη, ένα διάδρομο ενδεχομένω και με οικιανοκράνους για να γυρίσει ο κόσμος. Καλά, αυτό δεν είναι τώρα του παρόντος, ε, είναι το απότερου μέλλοντος θα ήταν ευχαρμόσυνο κάτι τέτοιο να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει, να υπάρξει κάποια ε, περιοχή ασφαλής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι πιθανό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθεί η διαδικασία Catch με τις αυθόρμητες τοποθετήσεις και έχω το πρόβλημα ότι έχουν ζητήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Δεν σας δώσω το λόγο σε όλους, γιατί δεν γίνεται, απλώς θα ήταν έφικτο. Η ώρα είναι ε, παρά έξι. Στις τέσσερις ακριβώς θα σταματήσουμε. Και αν δεν πάρετε το λόγο θα φτάνει οι προηγούμενοι συνάδελφοι που θα σας τον έχουν στερήσει. Γιατί θα έχουν μακρηγορήσει. Θυμίζω ότι έχετε ένα λεπτό για το ΚΑΤΣΔΙ. Η κυρία Πετήρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκπροσωπείται εδώ πέρα η οργάνωση Open Doors όπου έχουμε 10 χώρες όπου οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και η Συρία είναι πρώτη στον κατάλογο αυτών. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί σύντομα η κατάσταση και ότι θα αλλάξει αυτή η αντιχριστιανική